η διακοπή σαν την 12η Φεβρουαρίου ε, περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαναλαμβάνεται. Το πρακτικό και τα κείμενα που εγκρίθηκαν σε εκείνη την περίοδο συνόδου